Και το λόγο έχει ο κύριος Ριμπελίνη. Σενιόρ Ριμπελίνη, κύριε la palabra. Κύριε Ριμπελίνη, έχετε το λόγο. Δεν είστε, Ριμπελίνη. Κύριε Ριμπελίνη. Ο κύριος Μασίπ για ένα λεπτό. Ελπίζω τα δικήματα του κυρίου Μπελουσκόνη να διωχθούν από τη δικαιοσύνη και να σταματήσει η επικυριαρχία του στον τύπο. Μερικοί που δεν τον καταδίκασαν κάνουν τα στραβά μάτια. Αλλά αυτά που συμβαίνουν στην Ιταλία με τις ελευθερίες είναι πάρα πολύ σοβαρά και μας αφορούν όλους και ε, μας ε, απασχολούν όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μικεριτσιούτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα το σχέδιο ψηφίσματος ε, που συνέταξαν οι σοσιαλδημοκράτες με άλλες πολιτικές ομάδες διότι η ελευθερία έκφρασης, ε, πληροφόρησης ε, και διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να κατοχυρώνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι αυτό συνιστά θεμέλιο οποιασδήποτε ελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας. Η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προβλέπει ότι κάθε άτομο δικαιούται να εκφράζεται ελεύθερα και αυτή η ελευθερία έκφρασης καλύπτει την ελευθερία ελευθερία ελεύθερης τοποθέτησης χωρίς να παρεμβαίνουν οι δημόσιες αρχές. Οπότε οι βουλευτές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, και ανταγωνισμό μεταξύ τους σε εθνικό επίπεδο. Έτσι θα κατοχυρώσουμε την ελευθεροτυπία και οι δημόσιες αρχές ε, θα πρέπει να είναι σε θέση να την προστατεύσουν και να την προάγουν. Ε, αυτό συνιστά θεμελιώδη αρχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Βάγκελ για ένα λεπτό. Bien. Tiene la palabra por un minuto. Για ένα λεπτό τότε ο κύριος Μπελέτ. Ο κύριος Ριβελίνη, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Το τέλος του κόσμου φαίνεται να έφτασε για κάποιους, ενώ κάποιοι άλλοι βλέπουν ε, μια πεταλούδα να πετά. Κάποιοι λοιπόν βλέπουν τα πράγματα τελείως διαφορετικά και αυτό λέει ένας Κινέζος φιλόσοφος. Και εδώ το Νόμπελ Ειρήνης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την δήμωση του τύπου. Έχουμε το φαινόμενο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία και την ε, νοοτροπία του μίσους. Αυτό έδειξε η δημοσκόπηση αλλά αυτό έδειξε και η διαμαρτυρία για την ελευθερία του τύπου και η εικόνα του Πρωθυπουργού πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Διαμαρτυρία για την ελευθερία του τύπου στην Ιταλία. Θα πρέπει λοιπόν αυτό τον πολιτισμό του μίσους, τον αντιδημοκρατική επίθεση της, αριστερά, της αριστεράς των Ιακωβινιστών να την παρεμποδίσει το κοινοβούλιο μας. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αποφασιστικά να μην τα αναγνωρίσουμε όλα αυτά. Θα πρέπει η Ιταλία να μην καταντήσει η Ιταλίτσα. Ο Ιταλικός λαός δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο το μίσος της Ευρώπης να αλλάξουν τις διαστάσεις της χώρας. Ο πολιτισμός του μίσος, όποιος, ο πολιτισμός του μίσους δεν θα παρεμποδίσει την ε, δημοκρατική νίκη της κεντροδεξιάς στην Ιταλία να λάμψει. Κάποιοι αντιτίθενται στον κυβέρνηση, λίγοι είναι οι βουλευτές της κεντροαριστεράς, ακούγονται απόψεις όλων των ειδών, αλλά η αλήθεια έχει φτάσει στην αίθουσα αυτή. Πρέπει να περασπιστούμε τη δημοκρατία, πρέπει να συζητήσουμε και με την Ιταλική κεντροαριστερά που είναι ναρκωμένη, έχει πάρει ναρκωτικά και έχει την πολιτισμό του μίσους. Η κυρία Μορβάη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Στην Ουγγαρία ο κόσμος λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταπατάει τα δικαιώματα των πολιτών. Τελικά όμως ήταν η αποφασιστική η σημασία των τριών δεξιών Ούγγρων βουλευτών. Εμείς φροντίσαμε να μην περάσει το ε, ψήφισμα της αριστεράς. Δεν το λέω αυτό για λόγους κομματικής πειθαρχία, αλλά το οφείλουμε για λόγους ε, αλήθειας. Διπλά μέτρα και σταθμά δεν δεχόμαστε. Εχτες εκφράστηκαν παράπονα ενώπιον του Μπαρόσο ότι η σοσιαλφιλελεύθερη κυβέρνηση στην Ουγγαρία ε, δεν παραβιάζει την ελευθερία του τύπου. Μα οι άνθρωποι αυτοί πυροβολούν τον κόσμο στα μάτια, ε, συλλαμβάνει, ε, φυλακίζει, βασανίζει, κάνει εικονικές δίκες. Και μετά λέει ο Μπαρόσο αυτό είναι θέμα εσωτερικό της χώρας. Α ναι, και για την Ιταλία γιατί δεν είναι. Η δική μας αντιπροσωπεία δεν επιτρέπει τέτοια φαινόμενα καταπάτησης δικαιωμάτων. Για ένα λεπτό, η κυρία Ροντσούλη. Πρόεδρε, και πάλι ευχαριστώ. Η Ευρώπη καταγράφει ότι η Ιταλική αντιπολίτευση έχει περάσει σε μια παρεστησιογόνο κρίση θα προτιμούσαμε να μιλήσουμε για πραγματικά προβλήματα στην αίθουσα και να αναζητήσουμε και πραγματικές λύσεις. Τέλος πάντων μα παρηγορεί που η Ευρώπη καταλαβαίνει ότι μόνο ο κύριο Πιέτρο θα μπορούσε εδώ να θέσει ορισμένα θέματα προ τη ζήτηση. Από το 2004 πάντοτε με πρωταγωνιστή τον κύριο Πιέτρο παρασύρεται μια ολόκληρη μερίδα του Ιταλικού πολιτικού χώρου σε τέτοιε δράσει. Το ίδιο έγινε και εδώ σήμερα. Αυτή, αυτό το κίνημα λοιπόν, μεταξύ άλλων, φαίνεται ότι δεν πέτυχε, γιατί το Ιταλικό Εκλογικό Σώμα θέλησε να βγάλει από το σημερινό μας, ε, από το Κοινοβούλιο και τους κομμουνιστές που δεν παρίστανται στα έδρανα. Τώρα γίνεται επίθεση κατά του Πρωθυπουργού τη κυβέρνηση. Εδώ όμω δημιουργείται ένα κλίμα ανθρωποκυνηγητού, το οποίο επαναλαμβάνεται διαρκώ από την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Η κεντροαριστερά προκαλεί συνεχώ και αυτό έχει σοβαρότατε συνέπειε για όλου. Για ένα λεπτό, η κυρία Οντήρ. Πρόεδρε, ε, υπάρχουν μέσα για να καταστραφεί ο πλουραλισμό των μέσων μαζική ενημέρωση, για να μην υπάρχει ισορροπία στην παροχή ε, πληροφόρηση. Ε, υπάρχουν πολλά τέτοια μέσα για να συνθλίψουμε τις διαφορετικές απόψεις. Το μονοπόλιο στην πληροφόρηση μπορεί επίσης να επιτευχθεί όταν στην ηγεσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουμε μέλη της, ε, του κυβερνητικού σχηματισμού. Βλέπουμε πολλά γεγονότα που καταδεικνύουν ότι χρειαζόμαστε κανόνες πέρα από τον στόχο του να έχουμε μια ε, δημοκρατική Ευρώπη. Ε, χρειαζόμαστε μέσα για να προάγουμε τον πλουραλισμό και θα ήθελα να επικροτήσω τους παρασύνους για την πρότασή τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κασί για ένα λεπτό. Πρόεδρε, καταρχάς να διορθώσω την πρώτη και τη δεύτερη ψήφο μου. Ήθελα να απόσχω, αλλά έσφαλα διότι βιάστηκα και δεν χτύπησα το σωστό πλήκτρο. Μιλώ για τις πρώτες ψήφους της ημέρας. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με την αρχική πρωτοβουλία, ένα αμάρτημα που ήδη έχει εντοπίσει ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας σε σχέση με τη σημερινή πρωτοβουλία. Εδώ προστέθηκε η κίνηση της επίθεσης κατά του πρόεδρου της Ιταλικής Κυβέρνησης και η Ιταλική και η προσφυγή κατά των εφημερίδων του Ιταλικού τύπου. Εδώ για την πρωτοβουλία των διάφορων πολιτικών ομάδων ουσιαστικά δεν ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε για την πρωτοβουλία του ΕΛΚ. Μέτρα που διασφαλίζουν την Ιταλική αξιοπρέπεια, αφήνοντα όμω κατά μέρο τελείω το πρόβλημα ισορροπία μεταξύ κυβερνήσεων και αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και τύπου γενικότερα στι ευρωπαϊκέ χώρε, όχι μόνο στην Ιταλία. Η σύγκρουση συμφερόντων ε, δεν είναι μόνο περίπτωση που αφορά τον Ιταλό, Ιταλό Πρωθυπουργό. Το κόμμα μου λοιπόν αμφισβητεί την πλειοψηφία τη έγκριση του ψηφίσματο αυτού και εδώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα απέχοντα. Ευχαριστώ κύριε Καζίνη. Κύριε Σφιντάντσα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή αποδεικνύει ότι η Ιταλική αριστερά απέχει όλο και περισσότερο από το να ακούει την γνώμη του λαού μας. Εδώ δεν είχαμε συσπήρωση των Ιταλών, αλλά πολιτικό ελιγμό Και μια, έναν εκβιασμό πολιτικό των μέσων μαζικής ενημέρωσης του τύπου Κανείς δεν ξεχνάει ότι σήμερα οι Ιταλοί ανησυχούν για την ελευθερία του τύπου λόγω των κινήσεων του κυρίου Μπερλουσκόνη. Ο κάθε Ιταλός γνωρίζει ότι υπάρχουν εφημερίδες στην Ιταλία που ελέγχονται και έχουν όμως και άλλοι πολλοί μια γραμμή συντακτική που είναι αντίθετη από τον Ιταλό Πρωθυπουργό. Υπάρχει το μόνο αναγνωρισμένο σωματείο Ιταλών Πρωθυπουργών Ιτα... ε, αριστερής απόχρωσης. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Προσανατολισμός λοιπόν είναι απόλυτα αντίθετος με τον πρόεδρο της κυβέρνησης. Όλοι αυτοί εργάζονται και προχωρούν ανενόχλητοι στις εργασίες τους και ο πρόεδρος της κυβέρνησης ε, μάλλον δεν έχει απειλήσει κανέναν για την ελευθερία του. Εδώ υπάρχουν άλλα ζητήματα. Η κρίση, η λαθρομετανάστευση, η ανεργία, η συντάξη, αυτά είναι σοβαρά ζητήματα που θα έπρεπε να μα απασχολούν. Και όχι η αριστερά να ρίχνει αλλού το βάρο. Ευχαριστώ κύριε Καζίνη. Η κυρία Εκ παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα παραθέσω κάτι από τον Τζον Στιούρτ Μίλαν και μετά θα συνεχίσω στα Σουηδικά. Αν όλοι είχαμε μία άποψη, δεν δικαιολογείται η ανθρωπότητα να οδηγεί στη σύγχαση αυτού του ανθρώπου. Θα έπρεπε να σιωπήσει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Ε, λυπάμαι διότι έχει έτσι η κατάσταση σήμερα στην Ιταλία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να γίνει σεβαστή η ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τρόπο που ψηφίζει το ΕΛΚ δείχνει ότι αυτό δεν ισχύει ε, και ουσιαστικά κάνουν τι δουλειέ, ε, είναι παρατρεχάμενοι του Μπερλουσκόνη. Θα πρέπει να μην στερείται περιεχομένου το, το κράτος ε, για να γίνεται δημοκρατικός διάλογος ε, σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το πώς θα το πετύχουμε αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα, αλλά η κατοχύρωση της ελευθερίας είναι ευρωπαϊκό θέμα και λυπάμαι για την έκβαση της ψηφοφορίας για αυτό το ψήφισμα για την ελευθερία πληροφορίας στην Ιταλία. Ευχαριστούμε κυρία Εκ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, ο κύριος Μπερσκόν δεν με εντυπωσιάζει ούτε ηθικά ούτε πολιτικά και δεν είναι στο ζενήθ των κρατών με ελευθεροτυπία Ιταλία. Αλλά η ελευθεροτυπία και η ελευθερία της έκφρασης είναι κυρίως ζήτημα των Ιταλών, της Ιταλίας. Οι Ιταλοί οι ίδιοι να το ε, αναλάβουν. Και ευτυχώς αυτό συμβαίνει. Ε, ε κοιτάξτε τι γίνεται ε, με τις πρόσφατες εξελίξεις και η εφημερίδα Ελφάτο κοτιτιάνο δείχνει ότι υπάρχει και τύπος με κρίση και επικρίνει και λειτουργεί. Δεν υπάρχει θέμα λοιπόν και δεν νομίζω ότι θα πρέπει, ε, ούτε είναι ανάγκη να ασχοληθεί με αυτό η γραφειοκρατία των Βρυξελών. Εδώ δεν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, αλλά Ευρώπη που να προσανατολίζεται σε βασικές πυρηνικές αρμοδιότητες και μόνο τότε θα έχει την ε, εμπιστοσύνη των πολιτών η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριο Στάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι η ελευθερία πληροφόρησης είναι εξαιρετικά σημαντική και γι' αυτό ψήφισα έτσι. Αλλά, ξέρετε, συνεπάγεται και ευθύνες η ελευθερία στην ε, Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ε, ανοιχτή, διαφανή πληροφόρηση αλλά και επικριτική και θέλουμε να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Βλέπουμε στην ιστορία συγκεκριμένα παραδείγματα φημωμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης και ξέρουμε σε τι οδηγεί αυτό. Θα πρέπει ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσουμε σφαιρικά την κατάσταση στην Ένωση και όχι σε μία χώρα μόνο. Πρέπει να θεσπίσουμε αρχέ που θα ενστερνιστούμε όλοι, είτε μιλάμε για του ε, φιλελευθέρου, είτε μιλάμε για του σοσιαλδημοκράτες που είναι στην εξουσία. Πρέπει οι ίδιοι κανόνε να εφαρμόζονται για όλου, ε, και θα χρειαστεί να κατοχυρώσουμε την ελευθερία τη πληροφόρηση. Είναι μία από τι θεμελιώδει ελευθερίε, που ελπίζω θα, συνεχ... θα κατοχυρωθεί στην Ευρώπη και για το μέλλον. Ευχαριστώ κύριος Ντέιβις η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ε, λέει ότι εφαρμόζει ωραίες αξίες, ε, δημοκρατικές αξίες που κατοχυρώνονται μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, αλλά θέλω φλούμε σε αυτές τις κατάφορες παραβιάσεις που γίνονται σε κάποια κράτη-μέλη και δεν δαχτυλοδειχτούμε αυτούς που αποτυγχάνουν, δεν υποστηρίζουν τις αξίες στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σήμερα όμως την ευκαιρία να δείξουμε τι πιστεύουμε και να πούμε ότι ο έλεγχος των ε, ΜΜΕ από τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας συνιστά ε, σαφή παραβίαση. Υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα κράτη-μέλη. Απλά η χειρότερη κατάσταση σημειώνεται στην Ιταλία. Το UKIP ε, και οι συντηρητικοί έχασαν σήμερα με μία, μία ψήφο μόνο. Ο συντηρητισμό στη Βρετανία, το κίνημα, λέει ότι θα, πρέπει, θα θέλουν να εφαρμόσουν την κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λένε όμως ότι θέλουν να παρεμποδίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από το να αναλάβει οποιοδήποτε ρόλο και να υποστηρίξει τη δημοκρατία και τι θεμελιώδει αρχέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε τώρα για ένα λεπτό ο κύριο Κλάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που καταψηφίστηκε αυτό το ψήφισμα. Είναι απαράδεκτο το κοινοβούλιο αυτό να γίνεται αντικείμενο κατάκρισης για ε, πολιτική ε, αντίσταση κατά ενός πολιτικού θα γίνουμε ο μεγάλος αδελφός, ο ύψιστος ε, ιεροεξεταστής που ανακατευόμαστε σε θέματα που έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με τα κράτη-μέλη, το κάθε κράτος μέλος. Λεγόμενη απειλή κατά της πληροφορίας στην Ιταλία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εμείς είμαστε οι μόνοι ε, που είμαστε και οι πρώτοι κατάφυσης αριστερής υποκρισίας ε, που θέλει να ε, σκοτώσει έτσι τους πολιτικούς αντιπάλους. Και ε, αν ε, λυθούν τα πράγματα, προχωρήσουμε και στο Βέλιο και στην Ιταλία, θα έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάναν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δεν τιμάει το Κοινοβούλιο. Όλες οι ψηφοφορίες σήμερα, όλες οι ψηφοφορίες αφορούσαν ένα θέμα που ε, δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε ζητηθεί εδώ. Είναι εκτός των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου και είναι θέμα αποκλειστικό ενός κράτους μέλους. Εγώ δεν ε, αγαπώ ιδιαίτερα τον κύριο Μπερλουσκόνη και χαίρομαι που η Βρετανή Συνδυτική δεν είναι πια στο Λαϊκό Κόμμα. Αλλά είναι φαρισαϊκά αυτά που ακούμε ή αυτά ρέσκια της αριστεράς. Υποτίθεται ότι έχουν ασυλία, ε, ε, ε, αυτοί δεν έχουν ασυλία, ότι κυριαρχεί στον τύπο εκατοντάδες, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το κοινοβούλιο δαπανά στο να αυτοδιαφημίζεται και να αυτοπροβάλλεται. δεν είναι αυτό προ τιμήν ούτε των Ιταλών που έφεραν αυτό το θέμα εδώ και το έχασαν, ούτε τιμά εμά και του υπολείπου που είχαμε την ανέδεια να ανακατευτούμε σε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν εθνικοί μηχανισμοί δημοκρατικοί στο εσωτερικό τη Ιταλική Δημοκρατία. Και ε, ε, επαναλαμβάνω αυτό που λέω πάντα να θεθεί σε δημοψήφισμα η συνθήκη τη ότι θα πρέπει να ψηφιστεί. Ο κύριο Καμάλ έχει το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω όλοι σε αυτή την αίθουσα ενδιαφερόμαστε για την πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θέλουμε πάντοτε περισσότεροι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ανησυχώ για την πολυφωνία σε αρκετά κράτη-μέλη μεταξύ άλλων. Για την πολυφωνία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Όπου το θέμα αυτό δεν τίθεται καν, όπως στην Κούβα και την Βόρειο Κορέα. Εκεί να δούμε την πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως εδώ υπάρχει μια παταρχική αρχή Κάποιο είπε ότι δεν μπορούμε πάντοτε να έχουμε αυτό που θέλουμε. Όταν δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε αυτό που θέλουμε, πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε στη δημοκρατική διαδικασία των χωρών μα, ότι ο λαό έχει δικαίωμα να αντισταθεί στην κυβέρνηση όταν κάτι δεν το επιθυμεί. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να εγκρίνει δημοκρατικέ αποφάσει που όμω εκεί ανατρέπονται. Αυτή είναι η αρχή που οι συντηρητικοί υπερασπίζονται και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα υπερήφανο που η δική μα ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών καταψήφισε αυτό το αποτρόπαιο ψήφισμα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Σιλβέστρης. Πρόεδρε, νομίζω ότι η ψηφοφορία στην αίθουσα αυτή ε, τρόπο άριστο έδειξε δημοκρατικά την αλήθεια που όλοι γνωρίζουν ότι στην Αλία υπάρχει ελευθερία Ενημέρωση. Όμως η προσπάθεια τη αριστερά ήταν να εξεύρει επιχειρήματα για αντιπολίτευση γιατί στην Ιταλία, όπω έχουν πει πολλέ φορέ και άλλοι, υπάρχουν τόσε πολλέ εφημερίδες αλλά δεν ξέρουν τι γράφουν. Μπλοκάρουν, μπλοκάραμε τώρα για ένα μήνα τη δραστηριότητα της πρωτο, του κοινοβουλίου αυτού για να λέμε ότι στην Ιταλία δεν υπάρχει ελευθερία. Μα δεν γράφει πουθενά κάνει ότι η κυβέρνηση στην η Ιταλία στην ε, Καζεβέρ ε, με το σεισμό ανέλαβε αμέσω δράση ότι η νέα κυβέρνηση του Μπερλουσκόνη μάζεψε τα σκουπίδια από του δρόμου τη Νάπολη. Κανεί δεν το είπε από αυτό πουθενά. Λένε όμω οι εφημερίδε ότι η Ιταλία είναι μια χώρα όπου παρά την οικονομική κρίση Υπάρχουν τόσε θέσει εργασία. Το γράφουν αυτό στι εφημερίδε του. Γράφουν στι εφημερίδε του ότι παρά την οικονομική κρίση τράπεζε τη ε, Ιταλία είναι ε, ε, εύρωστε και έχουν χρήματα για του αποτομητευτέ. Κανεί δεν το λέει αυτό, κανεί δεν το γράφει και όταν το γράφουν το παίρνουν ω κοροϊδία και παραποίηση τη ελευθερία έκφραση. Στην Ιταλία λοιπόν υπάρχουν πολλοί που άνοιξαν το κουτί της παντόρας και προσπαθούν να βρουν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν και φήμωση τη δημοκρατία. Όμω η δημοκρατική διαδικασία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η ελευθερία στην έκφραση τη Ιταλία στην Ιταλία υπάρχει. Και όποιο ήθελε στην Ευρώπη να αποδείξει το αντίθετο απέτυχε. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε, για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την έκβαση τη ψηφοφορία για το ψήφισμα διότι η Ιταλία, κράτος μέλος της Ένωσης, και αναφέρεται με περιττό τρόπο μόνο αυτή μεμονωμένα σε μια πρόταση ψηφίσματο. Παρόλα αυτά πρέπει να συζητηθεί στο μέλλον η ελευθερία τη πληροφόρηση, η ελευθεροτυπία, η ελευθερία των δημοσιογράφων και των μέσων μαζική ενημέρωση για τα οποία δουλεύουν και για να το διασφαλίσουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και, ε, ε, αλλά σε ολόκληρη την Ένωση, όχι μόνο σε μία χώρα, θεωρούμε ότι σήμερα είναι με καλή μέρα για τη δημοκρατία και για την Ένωση. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό. Τελευταίος, ο κύριος Πατριτσέλα. Όπως λένε και αλλού, βρισκόμαστε στο Κοινοβούλιο και συζητάμε, ψηφίζουμε για ζητήματα που είναι περιτά και εδώ δεν ζητάμε, συζητάμε τις πρώτες προτεραιότητες που μας καίνε όλους. Την ε, πολιτική μετανάστευσης δεν συζητάμε και τις πρωτοβουλίες της Ιταλικής κυβέρνησης. Βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση εδώ προσπαθεί να αντιτεθεί στην ελεύθερη βούληση του λαού και φαίνεται να υπάρχει μια παράξενη συνωμοσία πολιτική, αλλά εδώ υπάρχει διαστρέβλωση και οργα... χειρο... χειραγώγηση της Ιταλικής πραγματικότητας με μόνο στόχο να καταστεί αναξιόπιστη κυβέρνηση Τη χώρα μας μέσω του προσώπου του Πρόεδρου τη του κυρίου Μπερλουσκόνη. Προσπάθηκαν κάποιοι να εκμεταλλευτούν εκλογικά και να κάνουν διαφημιστική εκστρατεία για ιδεολογικού σκοπούς, με ιδεολογικά επιχειρήματα και η εκστρατεία στρεφόταν ε, συστηματικά κατά συγκεκριμένων προσώπων, δίνοντα μια κακή εικόνα για τη χώρα μα στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν η Ιταλική αντιπολίτευση να συγκεντρωθεί σε ζητήματα που έχουν ε, πραγματικό, πραγματική σημασία για το κράτος, το ίδιο και η αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο, ζητήματα που έχουν ε, σημασία για τους πολίτες και να αφήσουμε κατά μέρο τι πρωτοβουλίε ενό κόμματο που συστηματικά εδώ και χρόνια επιτίθεται κατά του προσώπου του Προέδρου τη κυβέρνηση, που έχει εκλεγεί δημοκρατικά από 17 εκατομμύρια πολίτε. Ευχαριστώ κύριε Πατριτσέλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3.